Επαναλαμβάνεται η διακοπή στη συνεδρίαση. Τα χθεσινά συνοπτικά πρακτικά και τα κείμενα που εγκρίθηκαν διατίθενται. Έχετε αντιρρήσεις? Όχι από ό,τι φαίνεται. Ούτως λοιπόν εγκρίνονται